Dear Αγαπητοί συνάδελφοι, ας αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Σημείο 1 της ημερήσιας διάταξης, έγκριση της ημερήσιας διάταξης, τα σημεία 9, 14, 15 και 17 θα τα εξετάσουμε μετά το σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Τα δε σημεία 16 και 18 θα εξεταστούν μετά το σημείο 17. Τα σημεία 12 και 13 θα εξεταστούν μετά το σημείο 10. Τα σημεία 25 και 35 θα τα αναλύσουμε μετά το σημείο 11 της ημερήσιας διάταξης και τα σημεία 5, 7 και 26 αναβάλλονται. Μετά από έτοιμα του εισηγητή, σας προτείνω να συμπεριλάβουμε στα διάφορα το νέο σημείο εξέταση σχεδίου έκθεσης όσον αφορά τη συνθήκη του Μαρακέσα. Θα το εξετάσουμε αυτό μετά τα σημεία τα οποία θα εξεταστούν και κλεισμένων των θυρών. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποιες αντιρρήσεις ή παρατηρήσει, δεν νομίζω. Εγκρίνεται λοιπόν η παρατηρησει δεν νομιζω διάταξη, σημείο 2. ανακοινώσει του Πρόεδρου. Σα πενθυμίζω ότι ε, το εργαστήρι μα για την εφαρμογή τη οδηγία για τη διαμεσολάβηση θα λάβει χώρα αύριο στι 4.30 ε, το απόγευμα σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Θα ήθελα επίσης ε, ολόθερμα να σας προσκαλέσω στη δεξίωση που θα διοργανώσουμε προκειμένου να σηματοδοτήσουμε το ίμιση της εκλογικής αυτής ε, θητείας, της κοινοβουλευτικής συγχωρείτε θητείας, καθώς επίσης και την έναρξη της εορταστικής περίοδου. δεξίωση αυτή θα λάβει χώρα σήμερα στις 6.30, από τις 6.30 μάλλον και μετά, στην αίθουσα ASP 0G. Σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης, έγκριση των πρακτικών. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις και αν δεν λάβουμε ενστάσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, θα θεωρήσουμε ότι εγκρίναν τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 12ης και 13ης Οκτωβρίου. Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης, παρουσίαση της προσωρινής ερευνητικής εργασίας με θέμα πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα μοντέλο εγγύησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διάρκεια ζωής των προϊόντων. στο πλαίσιο της πρότασης οδηγίας για τις συμβάσεις όσον αφορά τις διαδικτυακές πωλήσει προϊόντων, η δική μας Επιτροπή ζήτησε την εκπόνηση μιας μελέτης, προκειμένου να ασχοληθούμε πιο συγκεκριμένα με το ζήτημα των προτύπων των μοντέλων εγγύησης για τη διάρκεια ζωής των προϊόντων. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω τον κύριο Κλάου Στόνερ, στον οποίο θα δώσω τώρα το λόγο, προκειμένου να μας παρουσιάσει εκ μέρους ερευνητικής ομάδας του Ινστιτούτου Διεν Finanzdienstlungen, το πόρισμα τη μελέτης αυτής που όπως σα είπα είχε το εξή θέμα, πώ θα μπορούσε να εφαρμοστεί στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα μοντέλο εγγύησης για τη διάρκεια ζωή των προϊόντων. Κύριε καθηγητά, έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σα για να κάνετε την παρουσίαση σα. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτέ, σα ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω ένα κομμάτι αυτής της πολύ σημαντικής έρευνας την οποία ζητήσατε και θα ήθελα να επικεντρωθώ στο ερώτημα πώς τα ζητήματα της ε, διάρκειας ζωής θα μπορούσαν να ρυθμιστούν νομικά από άποψη αστικού δικαίου. Αυτή τη στιγμή έχουν υποβληθεί δύο προτάσεις κομισιών που συσχετίζονται με αυτό το θέμα στενά και γι' αυτό δεν θέλω να επισέλθω σε γενικά ζητήματα που σχετίζονται με τη διάρκεια ζωής, αλλά με, να επισέλθω σε ε, συγκεκριμένα ζητήματα που σχετίζονται με αυτές τις δύο προτινόμενες οδηγίες. Under consideration αναφέρεται εδώ, ακριβώς γιατί δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα το έργο μας, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και φυσικά επιφυλασσόμαστε έως ε, το τέλος της ε, διάρκειας εκπόνησης της μελέτης μας να σκεφτούμε ενδεχομένως πράγματα που δεν έχουμε σκεφτεί ακόμη. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα σήμερα να σας παρουσιάσω μια πρώτη τάση που διαγράφεται. Το ε, σκεπτικό το οποίο θέλω να σας παρουσιάσω εδώ σε αυτά τα 10 λεπτά που έχω στη διάθεσή μου είναι ότι το ζήτημα της διάρκειας ζωής του προϊόντος δεν θα πρέπει να αφορά μόνο τον πολιτή αλλά και τον κατασκευαστή του προϊόντος. Βλέπετε εδώ στη διαφάνεια μία ε, σύνοψη ότι δεν μας ενδιαφέρει οποιοδήποτε κατασκευαστής, αλλά μόνο ο κατασκευαστής τεχνικών προϊόντων, ο οποίος Κατά τη δική μας γνώμη πιστεύει ότι θα πρέπει, πιστεύουμε μάλλον ότι θα πρέπει να ενημερώνει τους καταναλωτές για τη διάρκεια της ε, ε, ζωής του προϊόντος τους μέσω μιας commercial guarantee, μιας εμπορικής εγγύησης όπως ακριβώς ορίζεται στην οδηγία, την ισχύουσα οδηγία αλλά και στην πρόταση για την αγορά ε, ε επιγραμμικών προϊόντων με τη διαφορά ότι αυτή τη φορά θα πρέπει, θεωρούμε, να πρόκειται για δεσμευτική διάταξη. Ωστόσο, δεν θέλουμε να ορίσουμε υποχρεωτικές ελάχιστες διάρκειες ζωής, γιατί τα προϊόντα έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να ε, προσδιορίζονται για παράδειγμα δύο έτη διάρκεια ζωής, ελάχιστης διάρκεια ζωής για όλα τα προϊόντα. Αλλά πιστεύουμε ότι ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι ελεύθερος να ενημερώνει αν προσφέρει εγγύηση για τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, χωρίς να είναι υποχρεωμένος. Θα πρέπει όμως να αναφέρει ρητός ότι δεν το κάνει σε περίπτωση που πραγματικά δεν προσφέρει εγγύηση για τη διάρκεια ζωής. Γιατί επικεντρωνόμαστε στον κατασκευαστή. Πιστεύουμε ότι η ευθύνη του πολιτή δεν επαρκεί ακόμη και αν αντιστραφεί το βάρος της ε, υποχρέωσης ε, απόδειξης κατά την στη, χρονική στιγμή της παράδοσης του προϊόντος. Διότι δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο πολιτής ευθύνεται επί της ουσίας για την άριστη κατάσταση του προϊόντος κατά τη στιγμή της πώληση. Όχι παραπέρα. Ο πολιτής θα μπορούσε κανείς να πει ε, θα πρέπει να μπορεί να ε, αποδεικνύει την άριστη κατάσταση του προϊόντος του κατά τη στιγμή της πώληση. Ωστόσο, προφανώς, ε, κανείς δεν περιμένει ότι ένα μπουκέτο λουλούδια, για παράδειγμα, θα μπορούσε να διαρκέσει τρία χρόνια, να έχει διάρκεια ζωής, δηλαδή τρία χρόνια. Ποιος κατασκευαστής λοιπόν θα είναι. Δεν θέλουμε να επισέλθουμε στο δίκαιο για τα τρόφιμα ούτε να ε, ρυθμίσουμε τα ζητήματα των ανθόπολών. Θέλουμε να επικεντρωθούμε στα στους κατασκευαστές τεχνικών προϊόντων. Ποιος είναι αυτός, θα ρωτήσει ίσως κάποιος. Σας διαβεβαιώ ότι υπάρχουν πάρα πολλά νομοθετήματα τα οποία ορίζουν ακριβώς αυτό το θέμα. Εγώ πάντοτε ε, πάντοτε ε, παραπέμπω στην οδηγία ηλεκτρονικού και ε, ηλεκτρικού εξοπλισμού αλλά υπάρχουν και άλλες οδηγίες και κανονισμοί όπως για παράδειγμα η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό που αποσαφηνίζουν επαρκώς την, την έννοια του, κατασκευ... του κατασκευαστή τεχνικού προϊόντος. Δεν θέλουμε, όπως είπα, να προσδιορίσουμε ελάχιστη διάρκεια ζωής για όλα τα προϊόντα λόγω των μεγάλων διαφορών που χαρακτηρίζουν τα διάφορα προϊόντα. Θα μπορούσε βεβαίως κανείς να πει ότι θα μπορούσε να θεσπιστεί νομοθεσία κατά κατηγορία με, η οποία να ορίζει ελάχιστη διάρκεια ζωής των προϊόντων. Ωστόσο αυτό είναι κάτι που θεωρώ ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να το συζητήσουμε σήμερα μάλλον αφορά περισσότερο ε, ζητήματα που σχετίζονται με τα περιβαλλοντικά θέματα, τον οικολογικό σχεδιασμό κτλ. Εμείς ε, θα θέλαμε βεβαίως να συμβάλλουμε και σε εκείνη τη συζήτηση με βάση τη μελέτη που έχουμε εκπονήσει, αλλά δεν θα θέλαμε αυτή τη στιγμή να ε, προτείνουμε μια σειρά ε, μέτρων που θα πρέπει να ε, συζητηθούν στο πλαίσιο του οικολογικού σχεδιασμού. Σήμερα μιλούμε για το δίκαιο περιπολίσεων. Αν λοιπόν πρόκειται να θεσπιστεί νομοθεσία για αυτά τα θέματα, Πιστεύουμε ότι ο κατασκευαστής δεν θα πρέπει να είναι αλεύθερος απλά και μόνο για το ποια θα είναι η διάρκεια ζωής την οποία εγγυάται, αλλά θα ήθελα να θέσω ε, το εξή θέμα. Η διάρκεια ζωής δεν αφορά απαραίτητα και μόνο τον χρόνο. Θα μπορούσε κανείς να ορίσει χιλιόμετρα για παράδειγμα, τα οποία μπορεί να, διανύσει, ένα οχήματα ή πατήματα ενός κουμπιού για παράδειγμα, χρήσεις ενός πλυντηρίου. Θα μπορούσαν λοιπόν να ε, επιτρέπονται τέτοιου είδους περιορισμοί οι οποίοι θα πρέπει να διευκρινίζονται και να προσδιορίζονται από τον ίδιο τον κατασκευαστή και γι' αυτό κατά τη γνώμη μας η δική μας πρόταση είναι ε, φιλελεύθερη. Δεν προτείνουμε συγκεκριμένους περιορισμούς ε, ούτε συγκεκριμένες διατάξεις. Αντιθέτως ενθαρρύνουμε και παροτρύνουμε τους κατασκευαστείς τους κατασκευαστές προκειμένου να ορίζουν εκείνη το εύρος και τη διάρκεια αν θέλετε ή τον τρόπο με τον οποίο ε, ε, προορίζουν τα, τα προϊόντα τους για την χρήση. Δεν θέλουμε δηλαδή οπωσδήποτε ε, να επιτύχουμε τους σκοπούς που έχουν τεθεί μέσω απαγορεύσεων ή περιορισμών. Αν ωστόσο ε, ακολουθήσουμε μια τέτοια οδό, θα πρέπει κανείς να διαρωτηθεί πότε θα πρέπει να δίνονται αυτές οι πληροφορίες στους καταναλωτές. Εμείς λέμε στο σωστό χρόνο και στο σωστό τόπο. Και θέλουμε να συμπληρώσουμε την ομοθεσία που ισχύει ήδη. Μιλούμε πολύ συχνά και, και η Κομισιόν ε, το ίδιο το, για το ζήτημα της πλημμύρας πληροφοριών, άρα ζητούμενο είναι να ταξινομηθούν και να κατηγοριοποιηθούν με τέτοιον τρόπο οι πληροφορίες ώστε να είναι εύληπτες από τον καταναλωτή. Υπάρχουν και πολύ σημαντικές και πολύ ενδιαφέρουσες βέλτιστες πρακτικές. Θα μπορούσαμε για παράδειγμα να εμπνευστούμε από την οδηγία για την σήμανση των προϊόντων και θα πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι το μοντέλο με την εγγύηση του κατασκευαστή δεν αποτελεί μια απαλλαγή του πολιτή από τις δικές του ευθύνες. Αντιθέτως, αποτελεί ένα συμπλήρωμα και γι' αυτό θα πρέπει κατά την ενημέρωση του καταναλωτή να ε, παρέχεται ε, συγκεκριμένη αναφορά στο γεγονός ότι και ο πολιτής φέρει ορισμένες ευθύνες. Από αυτή την άποψη λοιπόν ε, η πρόταση που σας έχει υποβληθεί δεν αλλάζει κάτι. Παρ' όλα αυτά η πρόταση της Κομισιόν ε, θα ήταν κάπως ξεδοδιασμένη αν δεν προέβλεπε και κάποιες κυρώσεις και εδώ πιστεύουμε ε, βασιζόμενοι και στις ισχύουσες διατάξεις για τις εγγυήσεις ότι σε ορισμένες περιπτώσεις θα πρέπει να επιδιορθώνονται ή να αντικαθιστώνται τα, ε, προϊόντα εφόσον είναι ελοτηματικά και εφόσον δεν συμμορφώνονται και εφόσον ε, το αίτημα εγγύησης έχει υποβληθεί ε, του οριζόμενου χρόνου ή της οριζόμενης περίοδου από τον κατασκευαστή. Αν ωστόσο ο κατασκευαστής δεν αναλάβει καμία δράση, δηλαδή δεν συμπληρώνει το προϊόν του με, κάποιο, με κάποια πληροφορία και εκεί πιστεύουμε ότι θα πρέπει να επιβάλλεται κάποια κύρωση και σκεφτόμαστε αυτό, τον, ε, αυτό το διάστημα ε, μήπως θα έπρεπε ο, πολι, κατασκευαστής να, να ευθύνεται όπως και ο πολιτής. Τώρα, για τους ε, χρόνους παραγραφής για τους ε, πολιτές. Ένα λεπτό. Ε, μια πρόταση. Το πρόβλημα ε, στο ζήτημα της, ε, της παραγραφής θεωρούμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η αντιστροφή του, της υποχρέωσης απόδειξης ε, θα πρέπει να βαρύνει την ε, Κομισιόν. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω το σκεπτικό μας, αλλά αυτό που, που προτείνουμε είναι μια περίοδο 2 συν 2, 2 χρόνια εγγύηση, 2 χρόνια αντιστροφή απόδειξης, από ότι ε, την προτινόμενη διαδικασία του 3 συν 1. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί ακόμη όμως ε, πρέπει να σας πω. Ε, σας έδωσα μια παροκατακτική εικόνα για το πού κινείται η δική μας σκέψη. Αυτά από τη δική μου πλευρά. Αν δείτε και τις διαφάνειες, ε, εκεί υπάρχει και μια συγκεκριμένη πρόταση για τη διατύπωση που έχουμε κάνει, αλλά δεν θέλω να επισέλθω και να σας τη διαβάσω. Οπότε αυτά από μένα και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, καθηγητά Τόνερ, για την παρουσίαση αυτή. Να δώσω τώρα το λόγο στην εισηγήτρια, η οποία θα συντάξει μια γνωμοδότηση όσον αφορά την οδηγία για τις συμβάσεις διαδικτυακών πωλήσεων προϊόντων. Αναφέρομαι στην κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τον καθηγητή κύριο Τόνερ για την σημαντική αυτή παρουσίαση που έκανε. Πρέπει να δούμε όντως αν θα είναι ρεαλιστική μια τέτοια εγγύηση και αν θα μπορούσε να εφαρμοστεί στη διαδικτυακή πώληση προϊόντων. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να αναφερθώ σε συγκεκριμένα σημεία που έχουν να κάνουν με την εγγύηση αυτή και τη διάρκεια ζωής. Νομίζω κύριε καθηγητά ότι πραγματικά οριοθετήσατε πάρα πολύ καλά που βρίσκονται τα δικαιώματα, που οι υποχρεώσεις και που η ευθύνη που φέρουν τα συμβαλόμενα μέρη. Είναι ενδιαφέρουσα επίσης η προσέγγισή σας. Αν κατάλαβα καλά προσπαθείτε να συνδυάσετε από τη μια πλευρά μια εθελούσια προσέγγιση και από την άλλη όμως θέλετε να υπάρχουν και κάποιε κυρώσει οι οποίε αν κατάλαβα καλά θα πρέπει να λειτουργήσουν ενθαρρυντικά για τους παραγωγούς, για τους κατασκευαστές, να είναι υποχρεωτικό με λόγια για τον παραγωγό, να αναλαμβάνει τις ευθύνες του όσον αφορά τις ε, δεσμεύσεις τελικά που παίρνει με την κατασκευή ενός προϊόντος. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω λίγο περισσότερο την προσέγγιση αυτή. Πολύ συχνά έχουμε αναφερθεί στην εθελούσια προσέγγιση και προσπαθούμε να τη συνδυάσουμε κάποιου δεσμευτικού κανόνε. Ενδεχομένω λοιπόν η δική σου προσέγγιση ήταν και πιο καινοτόμα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, αναφερθήκατε στην παρουσίασή σα σε διάφορα νομοθετικά μέσα τη κοινότητα τα οποία έχουν κοινά χαρακτηριστικά, θα έλεγα, κοινού ε, κανόνες ε, σε σχέση με την διάρκεια ζωής ε, των προϊόντων. Ίσως λοιπόν θα μπορούσατε να μας δώσετε λίγο περισσότερες εξηγήσεις για το πώς μπορούμε να εντοπίσουμε καλύτερα τα νομοθετικά αυτά μέσα, πώς τα επιλέξατε, και πώς τελικά καταλήξατε να προτείνετε αυτό το οποίο ενδεχομένως θα προτείνετε τελικά στη μελλοντική σας μελέτη. Και τέλος, μου ακούγεται απόλυτα λογικό αυτό το οποίο είπατε, ευθύνη των παραγωγών, των κατασκευαστών συγκεκριμένων τεχνικών προϊόντων, που όπως εξηγήσατε προφανώς δεν μπορούμε να αναφερθούμε εδώ πέρα σε αγροτικά προϊόντα, αναφερθήκατε σε λουλούδια για παράδειγμα, σε άνθη, Προφανώς δεν θα μπορούσαμε να τα καλύψουμε από τέτοιε ε, τεχνικές προδιαγραφέ. Πώς γίνεται λοιπόν να έχουμε μια κοινοτική νομοθεσία η οποία θα μπορούσε να μας οδηγήσει στον απότερο στόχο μας, ε, μια εκτεταμένη διάρκεια ζωής των προϊόντων, η οποία να αποτελεί μια μορφή υποχρέωσης, αν θέλετε, για τους κατασκευαστές. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει και εμείς να προωθήσουμε ως νομοθέτες. Ζούμε σε έναν κόσμο που σπαταλά και εξαντλεί πολλές φορές τους φυσικούς του πόρους. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να νομοθετήσουμε υπέρ της βιωσιμότητος και της διάρκειας ζωής των προϊόντων. Νομίζω ότι ορισμένοι έχουν πει ότι πολλές φορές καταναλώνουμε το αντίστοιχο πολλών διαφορετικών πλανητών όσον αφορά το μέγεθος των πόρων που καταναλώνουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αλλάξουμε ρότα και εμεί ως νομοθέτε να καταφέρουμε να πείσουμε του παραγωγού, κατασκευαστέ ότι θα πρέπει να ακολουθούν διαφορετική προσέγγιση. Νομίζω ότι όλα αυτά τα σημεία θα πρέπει να εμπνεύσουν τι συζητήσει που θα κάνουμε όσον αφορά τη διάρκεια ζωή των τεχνικών αυτών προϊόντων. Τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Άρημον, το οποίο είναι ο συλληγητής στην καθήλυνα αρμόδια επιτροπή την ΙΜΚΟ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να επισημάνω ότι θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τόνερ για αυτήν την ε, γνωμοδότηση την οποία και έλαβα 16 ή 17 Νοεμβρίου διότι ε, με επισκέφτηκε η Οργάνωση Καταναλωτών της Γερμανίας ε, συζητήσαμε λοιπόν αυτό το θέμα και με βάση τις ιδέες που εκφράστηκαν, ε, μπορώ να σας πω ότι έκανα πολλή δουλειά. Γιατί ασχολήθηκα εντατικά με το πώς θα μπορούσαμε να εντάξουμε αυτό το ζήτημα της διάρκειας ζωής των προϊόντων σε ένα νομοθετικό κείμενο, χωρίς όμως να δημιουργούμε μια γκρίζα νομική ζώνη, η οποία να επιτρέπει τη διαφορετική αξιολόγηση κάθε προϊόντος προκειμένου να μην χρειάζεται δηλαδή σε κάθε αγορά ο καταναλωτής να πρέπει να ανατρέχει σε κάποιον κατάλογο προκειμένου να διαπιστώνει πόσο, πόση θα είναι η εγγυημένη διάρκεια ζωής του. Το ίδιο λένε και πολλές επιχειρηματικές ενώσεις ότι ένα τέτοιο μοντέλο θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα εφαρμόσιμο και δεν θα πρόσφερε ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τις εγγύησεις. Θα ήταν δε και πάρα πολύ περίπλοκο να θέσει κανείς ένα τέτοιο σύστημα σε εφαρμογή σε μια ενιαία αγορά. Θεωρώ λοιπόν ότι η ιδέα σας ότι αυτό δεν θα έπρεπε να ρυθμίζεται νομοθετικά από τα πάνω, δηλαδή από το κράτος, αλλά ότι καλύτερο θα ήταν αυτή η διάρκεια ζωής να καθορίζεται στο επίπεδο του κατασκευαστή. Την αποδέχομαι αυτήν την ε, ιδέα και τη θεωρώ και πολύ ενδιαφέρουσα, ιδίως και στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και ιδίως και στο πλαίσιο ότι οι κατασκευαστές θα πρέπει να σχεδιάζουν τα προϊόντα τους με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορούν να τίθενται σε χρήση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Πολύ δύσκολο ε, λοιπόν είναι το, το ζήτημα που αφορά την διάρκεια ζωής ενός προϊόντος, ακριβώς γιατί δεν είναι πάντοτε η ίδια. Ε, είναι άλλο θέμα όταν κάποιος χρησιμοποιεί, για παράδειγμα, η συχνότητα δηλαδή της χρήσης ε- ενός προϊόντος επηρεάζει και την ε, διάρκεια ζωής του, προϊόντο. του προϊόντος. Ίσως αυτή η ιδέα σας λοιπόν ότι η ελάχιστη διάρκεια ζωής δεν θα πρέπει να αφορά μόνο τον χρόνο, αλλά ενδεχομένως και τον αριθμό των χρήσεων, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Είπατε επίσης ότι όλοι εκείνοι οι κατασκευαστές που δεν ε, προσφέρουν κάποια εγγύηση για τη διάρκεια ζωής του προϊόντος τους, θα πρέπει να εξισώνονται με τους πολιτές και να, να λαμβάνουν και εκείνοι ένα μέρος της ευθύνης. Ένα ερώτημα. Αυτό σημαίνει ότι αυτό που στο, στη βελγική νομοθεσία αναφέρεται ως ε, αξιών direct, ε, την, ε, την ε, δυνατότητα δηλαδή του καταναλωτή να μην προσφεύγει μόνο κατά του, καταναλω... του πολιτή αλλά και του κατασκευαστή ενός προϊόντος. Εγώ βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα αυτή την ιδέα και είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολλές επιλογές. Έχετε ελέγξει ε, τι συμβαίνει, τι θα συμβαίνει ε, στις περιπτώσεις όπου ένας κατασκευαστής δεν γράφει μεν μηδέν πάνω στο προϊόν, στο προϊόν του, αλλά που, το, που ο κατασκευαστής ορίζει μια διάρκεια ζωής η οποία είναι χαμηλότερη από την νομικά προβλεπόμενη. Μήπως θα, θα έπρεπε δηλαδή με κάποιον τρόπο να υποχρεώνονται οι κατασκευαστές να προσφέρουν εγγύηση ίση ή τουλάχιστον ίση με εκείνη που προβλέπεται στην νομοθεσία. Και τι θα συμβαίνει, αυτό είναι το ερώτημά μου, ε, σε περίπτωση που ένας κατασκευαστής ορίζει εγγύηση για τη διάρκεια ζωής χαμηλότερη από εκείνη που προβλέπει η νομοθεσία. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα που συνδέεται με το πρώτο μου είναι αυτό το πολύ κρίσιμο ζήτημα της ε, αντιστροφής της ε, ε, απόδειξης είναι πολύ περίπλοκο το θέμα αυτό. Προς το παρόν η Κομισιόν προτείνει μια περίοδο δύο ετών, αλλά και εδώ το ερώτημά μου είναι πώς θα μπορούσαν αυτές οι προθεσμίες, αυτές οι διορίες να ενοποιηθούν με έναν τρόπο ώστε να υπάρχει μια συνοχή. Γιατί είναι δύσκολο και για τον καταναλωτή αλλά και για, τον κατασκευαστή να αναλάβει ε, την ευθύνη απόδειξης. Ε, ε, άρα πρέπει να βρούμε ποια, με ποιον τρόπο θα ρυθμιστεί αυτό το θέμα. Σε ένα αυτοκίνητο, για παράδειγμα, θα ορίσουμε 200.000 χιλιόμετρα, 150.000 χιλιόμετρα, 4-5 χρόνια. Ε, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ρυθμίσουμε και αυτό το ζήτημα που, που αφορά την διάρκεια ζωής του προϊόντος. Ο κύριος Φως. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τόνερ για την παρουσίασή σας και για την ε, για τις ιδέες σας. Εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός όταν ακούω να, ε, να παρέχονται διαρκώς νέες ε, πληροφορίες στον καταναλωτή. Ε, κάτι που ενδεχομένως θα δυσκολέψει και τους κατασκευαστές στις δραστηριότητες τους, χωρίς ωστόσο να προσφέρει κάποιο όφελος για τον καταναλωτή. Ε, γιατί στην ουσία υπερφορτώνεται με πληροφορίες. Παρ' όλα αυτά θέλω να δείξω ότι είμαι καλός μαθητής. Και θα ήθελα γι' αυτό το λόγο να σας κάνω κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις για να κατανοήσω καλύτερα αυτά που είπατε. Θεωρείτε λοιπόν ότι όταν αναφέρει ένας κατασκευαστής μια ημερομηνία ή μια διάρκεια ζωής, και δεσμεύεται από αυτήν. Αυτό όμως αντίστροφα δεν θα σημαίνει ότι και το εκάστοτε προϊόν θα γίνεται ακριβότερο για τον τελικό καταναλωτή. Δεν θα πρέπει αυτό το κόστος να μετακυληθεί στην τιμή του προϊόντος. Μήπως λοιπόν οι πολίτες μας τελικά θα καταλήξουν να πληρώνουν περισσότερα χρήματα προκειμένου να λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες που εσείς προτείνετε. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Δεύτερον, πόσο μεγάλο θα είναι το βάρος ε, για τις επιχειρήσεις. Ε, πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό που προτείνατε. Ας σκεφτούμε μια γόμα. Στα τρόφιμα τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Προφανώς τα, πράγματα, τα τρόφιμα κάποια στιγμή έχουν μια ημερομηνία λήξης και λήγουν. Τι θα γίνει όμως σε μια γόμα για παράδειγμα ή σε ένα μολύβι. Αυτό εξαρτάται από τη χρήση που θα του κάνει ο καταναλωτής. Πώς θα μπορούσε ένας κατασκευαστής να ορίσει ποια είναι η διάρκεια ζωής αυτού του προϊόντος. Στα, στα χαλιά για παράδειγμα. Θα πρέπει ε, ο κατασκευαστής να, να καθορίσει πόσα άτομα θα περπατούν κάθε μέρα πάνω σε αυτό το χαλί. Ε, αλλά ε, όταν είναι να αγοράσω ένα χαλί για το σπίτι μου, ε, προφανώς τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά ή ξέρω εγώ για παράδειγμα σε, σε, σε ένα καλάθι ε, που μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί μηχανικά για να ανεβοκατεβάζει πράγματα εξαρτάται πόσες φορές και τι είδους αντικείμενα θα τοποθετεί μέσα σε αυτό το καλάθι. Το ίδιο Θέλω να πω, σε μια μπαταρία τα πράγματα μπορεί να είναι κάπως πιο ξεκάθαρα, αλλά πάντοτε ε, επηρεάζονται τα πράγματα και από την χρήση, από την συχνότητα της χρήσης, την ένταση της χρήσης. Ε, δεν ξέρω, ε, σας θέτω όλα αυτά τα ερωτήματα για να μπορέσω να καταλάβω λίγο καλύτερα αυτά που μας είπατε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκέπαρτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Τόνερ για αυτήν, την, αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες που μας παρουσιάσατε. Πιστεύω ότι ε, την ε, εποχή της ψηφιοποίησης ε, την οποία διανύουμε είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό να καινοτομούμε και στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών χωρίς να χρησιμοποιούμε πάντοτε τις πεπατημένες που μιλούν για εγγυήσεις, για εχέγγυα κτλ. κτλ. Γνωρίζουμε ότι πολλά πράγματα σήμερα δεν λειτουργούν γιατί ε, στους κανόνες, ε, στην νομοθεσία ακριβώς προβλέπονται οι ίδιες μάλλον προθεσμίες ε, για προϊόντα που κυμαίνονται από μια γόμα μέχρι ένα αυτοκίνητο. Αλλά θα ήθελα πραγματικά το αυτοκίνητό μου να διαρκέσει λίγο πιο πολύ από ότι το μολύβι που θα αγοράσω. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η καινοτομία που κομίζετε εσείς με τις προτάσεις σας Και αν κατάλαβα καλά, κύριε Τόνερ, μιλάτε για μια υποχρέωση ενημέρωσης του κατασκευαστή. Δηλαδή ο κατασκευαστής θα είναι υποχρεωμένος να παρέχει ορισμένες μια πληροφορία η οποία όμως θα μπορούσε να είναι και μηδέν, να είναι μηδενική, ότι δεν προσφέρει εγγύηση καθόλου. Απλά θα καλεί το ίδιος ο κατασκευαστής να ορίζει ποια πιστεύει ο ίδιος ότι θα πρέπει να είναι, ότι θα είναι η διάρκεια ζωής του προϊόντος που κατασκευάζει. Ε, εγώ πολύ συχνά ε, στα καταστήματα ε, στα οποία αγοράζω τα προϊόντα μου μου μου προσφέρονται πρόσθετες εγγύησεις. για, το αυτοκίνητό μου, για παράδειγμα, αγόρασα συν πέντε χρόνια εγγύηση. Ε, αυτά θεωρώ ε, ότι ίσως και αυτό θα ήταν μια ενδιαφέρουσα ιδέα. Πολύ ενδιαφέρουσες οι ιδέες σας πάντως σε κάθε περίπτωση, γιατί θα μπορούσαν να αποτελέσουν και μια παρότρινση προς τους κατασκευαστές, προκειμένου να προσεγγίσουν και με έναν νέο, με έναν καινοτόμο τρόπο ε, τα δικά τους προϊόντα, όχι μόνο στο σχεδιαστικό κομμάτι, αλλά και στο τεχνικό καθαρά κομμάτι. Γιατί πολλές φορές έχουμε την αίσθηση ότι ε, κάποια προϊόντα φαίνεται σαν να έχουν μια κρυμμένη ημερομηνία λήξης. Βέβαια, τίθεται πράγματι το ερώτημα. Σε περίπτωση που προβλέπετε μια ελάχιστη διάρκεια ζωής ε, δύο ετών, το οποίο αποτελεί ελάχιστο κανόνα, Θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να τροποποιηθεί αυτό. Και κάποιος κατασκευαστής στη συνέχεια πει ότι ε, το πλυντήριό μου έχει εγγύηση για ένα χρόνο ή για ενάμιση χρόνο. Δεν υπάρχει ένας κίνδυνος εδώ να προσφέρονται ε, ε, αντιφατικές πληροφορίες Όσον αφορά την αντιστροφή της απόδειξης, συγγνώμη κύριε Αρημό, αλλά εγώ πιστεύω ότι ο κατασκευαστής είναι πολύ πιο εύκολο να αποδεικνύει πού και για ποιο λόγο εμφανίστηκε κάποιο ελάττωμα στο, προϊό, προϊόν του, από ότι ο καταναλωτής, ο οποίος το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να χρησιμοποιήσει το προϊόν που έχει αγοράσει. Γι' αυτό θεωρώ ότι αυτή η αντιστροφή της υποχρέωσης απόδειξης ε, ε είναι ε, σωστή ε, προσέγγιση, γιατί εκείνος που μπορεί να αποδείξει και που έχει τα μέσα για να περάσει σε μια τέτοια απόδειξη, θα πρέπει να είναι και εκείνος που θα υποχρεούται να το κάνει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Οι, οι διαφορές που υπάρχουν σε αυτές τις συμβάσεις ε, είναι πολύ σημαντικές και αφορούν το διασυνοριακό εμπόριο όλες οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να ε, αναλαμβάνουν ε, επιπρόσθετο κόστος, επιπρόσθετες δαπάνες. Η ενιαία αγορά απαιτεί ενιαίες ρυθμίσεις ε, για όλες τις εξαποστάσεις πωλήσει τις επιγραμμικές. Η διαφορά στους ρυθμίσεις και στους κανόνες στις πωλήσει μέσω διαδικτύου οδηγεί σε κατακαιρματισμό. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά αυτές τις προκλήσεις. Πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες δεν ψωνίζουν διαδικτυακά διότι δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ανησυχούν να προβούν σε αυτές τις αγορές. Χρειαζόμαστε λοιπόν γενικούς κανόνες που αφορούν στην προστασία των καταναλωτών, μια απόλυτη εναρμόνιση θα επιτρέψει την βελτίωση της προστασίας ε, στα κράτη-μέλη της Ένωσης. Και αυτό θα αποτελούσε μια σημαντική επιτυχία. Θα πρέπει να βρούμε επίσης ε, λύσεις που να αφορούν και τα υπόλοιπα κράτη, κάτι το οποίο θα διευκολύνει την πρόσβαση των ε, καταναλωτών στις αγορές τις διαδικτυακές. Θα πρέπει να πετύχουμε μια ισορροπία και δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται περαιτέρω οι επιχειρήσει. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάπτα λέει το λόγο. Ευχαριστώ. Φυσικά όλοι θέλουμε να μάθουμε ποια είναι τα προϊόντα τα οποία μπορούν να εντοχθούν σε αυτήν την, ε, οργανισμό, σε αυτή την ε, οδηγία. Και ε, τώρα οι διαδικασίες ε, ελέγχου, τεσταρίσματος, ε, να αγοράσουμε κάποια έπιπλα και μερικές φορές ο <clears throat> πολιτής λέει ότι ένας, ένα σκύλο μπορεί να χορπηδήσει σε αυτό τον καναπέ και στο ύφασμα που τον καλύπτει 100.000 φορές. Πώς μπορούμε λοιπόν να επαληθεύσουμε αυτές τις ε, εγγύησεις ε, για όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Ο απογοητευμένος ε, αγοραστής, καταναλωτής, πώς μπορεί να αποδείξει ότι το σκυλάκι χοροπήδησε λιγότερο από 100.000 φορές και ο καναπές έσπασε. Ευχαριστώ κύριε Άντερσον. Δεν είμαι μέλος της Επιτροπής σας, Είμαι σκιώδης των σοσιαλιστών ε, πάνω στο θέμα και νομίζω ότι τα σχόλια που έκανε η Εύελιν ε, ειδικά είναι πολύ σωστά. Η ιδέα αυτή είναι καλή, αλλά όλοι γνωρίζουμε στην ουσία ότι σε πολλές περιπτώσεις οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν τα εγγυήσεις και τα δικαιώματά τους. Και όταν η περίοδος εγγυήσεις έχει παρέλθει, θα πρέπει να παραιτηθούν και να δεχθούν ότι το προϊόν χάλασε, είτε πρόκειται για έναν φορητό υπολογιστή, είτε για ένα πλυντήριο. Πέρασε η περίοδο εγγύηση και δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Ακόμα και αν ε, έχουν δικαίωμα, τώρα εξάρτητα από την αντιστροφή του βάρου απόδειξη, υπάρχουν καλά προβλήματα, διότι ε, υπάρχουν, υπάρχουν κατασκευαστέ, όχι καλοί κατασκευαστές δεν καθιστούν σαφώς, σαφές στους αγοραστές ότι έχουν δικαιώματα και μετά από το ε, παρέλευση ενός, δύο ή τριών ετών εγγύησης. Λοιπόν, κάτι στο οποίο θα δίνουν περισσότερες προφορίες είναι μια πολύ καλή ιδέα και συμφωνώ ότι θα πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα πρέπει να αφαιθεί στην καλή πρακτική, την πρακτική ή την βιομηχανική πρακτική. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να συμπεριληφθούν σε μια οδηγία. Επίσης ε, καλωσορίζω τα σχόλια τα οποία κάνουν διάκριση ανάμεσα στον, ε, ε, στην νο, περίοδο διάρκειας και την περίοδο της εγγύησης, διότι το θέμα της διάρκειας εγγύησης, διάρκειας εγγύησης είναι όντως κάτι το οποίο περιορίζει σε κάποιες περιπτώσεις. Και, αλλά δεν είναι σωστό διότι Ε, αν χρειαστεί να εφαρμόσουμε αυτή την ζωφή του βάρους απόδειξης, τότε θα θέλαμε να ακούσουμε κάτι παραπάνω πάνω στο θέμα. Ευχαριστώ. Κυρίως ως ε, τον ΕΡ θα απαντήσει. Φυσικά ε, συζητάμε ένα ενδιάμεσο έγγραφο. Θα βρούμε τις απαντήσεις στο τελικό έγγραφο Παρακαλώ απαντήστε κύριε καθηγητά σε ό,τι μπορείτε, αλλά όχι ε, αναλυτικά σε όλες τις ερωτήσεις, γιατί δεν έχουμε τον επαρκή χρόνο. Ευχαριστώ. Ομολογώ ότι ο κύριος Αριμό ε, επισήμανε ένα πολύ προβληματικό ε, θέμα. Φυσικά, κανένας κατασκευαστής δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να μπορεί να προσφέρει μικρότερη εγγύηση από αυτή που προσφέρει ο, ε, που προβλέπει ο νόμος. Άλλωστε υπάρχει ήδη ε, σχετική διάταξη στην νομοθεσία και γι' αυτό το λόγο πιστεύουμε ότι θα πρέπει να καταστεί πιο σαφής και πιο αυστηρή ε, η συγκεκριμένη διάταξη. Προ το παρόν δεν έχω απάντηση στο ερώτημά σας, το εξετάζουμε ακόμη. Όσον αφορά την αντιστροφή του βάρους απόδειξη, εμείς πιστεύουμε ότι ε, θα πρέπει, ε, όπως προτείνει και η Κομισιόν, να συνδυάζεται με την παροχή εγγύησης, χωρίς ωστόσο να θεωρούμε ότι είναι πανάκια. Ο ε, ο πολιτής σε ορισμένες ε, περιπτώσεις μπορεί ε, πράγματι να σε ορισμένες περιπτώσεις να καλύπτεται από την ισχύουσα νομοθεσία όπως σε αναλώσιμα ή σε λουλούδια όπως ανέφερα νωρίτερα. Κύριε Φως, θέσατε το ερώτημα μήπως ε, αυξηθεί το κόστος των προϊόντων με αυτόν τον τρόπο. Εγώ ε, ε, είμαι πολύ προσεκτικός ως προς τις λύσεις που προτείνω και αναφέρω ρητός αυτό που δεν θέλω σε καμία περίπτωση είναι μέσω τέτοιων νομοθετικών διατάξεων να αναγκαστεί ο κατασκευαστής να ορίσει συγκεκριμένη διάρκεια ζωής. Ας πάρουμε το παράδειγμα με το πλυντήριο. Ο καταναλωτής πιστεύω ότι θα πρέπει και μετά τη θέσπιση μιας τέτοιας διάταξης να ε, ε, έχει την επιλογή αν θα αγοράσει ένα φτηνό πλυντήριο που βεβαίως θα του κρατήσει μόνο τρία χρόνια ή αν θα αγοράσει ε, ένα ακριβότερο πλυντήριο το οποίο όμως θα το έχει στη διάθεσή του για περισσότερα χρόνια. Αυτή την επιλογή δεν θέλουμε να του την αφαιρέσουμε του καταναλωτή αλλά θα πρέπει να είναι ενήμερος εκ των προτέρων κατά τη στιγμή της αγοράς του και νομίζω ότι από αυτή την άποψη κάτι τέτοιο θα ήταν το ιδανικότερο. Είναι λοιπόν μια πρόταση η οποία σέβεται την οικονομία της αγοράς. Όσον αφορά τις ε, προθεσμίες ε, για την ε, παροχή εγγύησης, περιμένουμε ακόμα ορισμένες πληροφορίες από εμπειρογνώμονες στα διάφορα κράτη-μέλη. Έχουμε ήδη λάβει κάποιες απαντήσεις, χωρίς ωστόσο να έχουμε καταφέρει να αξιολογήσουμε όλα τα στοιχεία μέχρι στιγμής. Όταν λάβουμε όλα τα στοιχεία και λάβουμε και τις ε, πληροφορίες από κράτη-μέλη τα οποία έχουν ορίσει στη δική τους νομοθεσία μεγαλύτερη ε, εγγύηση ε, πώς αποφεύγουν εκείνα τα κράτη-μέλη το πρόβλημα της παραγραφής της ευθύνης. Αυτό είναι κάτι που πράγματι λείπει αυτή τη στιγμή από τη δική μας πρόταση. Και ως προς το ζήτημα των τεχνικών προϊόντων επίσης είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί θέλουμε σε πρώτη φάση να επικεντρωθούμε στα τεχνικά, ε, στα τεχνικά προϊόντα και μόνο. Εσείς αναφερθήκατε και σε μια άλλη κατηγορία ή σε άλλες κατηγορίες προϊόντων, όπως για παράδειγμα τα έπιπλα. Θα πρέπει βεβαίως να σκεφτούμε και σε αυτές τις περιπτώσεις τι θα πρέπει να γίνει, αλλά θεωρούμε ότι σε επίπεδο ενωσιακής νομοθεσίας θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια πολύ προσεκτική και αργή, θα μου επιτρέψετε να πω, βαθμιαία προσέγγιση, ακριβώς γιατί... Ε, ε τα θέματα αυτά είναι ε, καινούρια, είναι και αχαρτογράφητα ύδατα και θεωρούμε ότι τα τεχνικά προϊόντα είναι ένας τομέας όπου μπορούν πραγματικά να γίνουν κάποιες πρώτες δοκιμές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τόνερ. Αυτά είχατε να ε, πείτε ως απάντηση ε, από ό,τι καταλαβαίνω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ και αναμένουμε την παρουσίαση του τελικού ε, εγγράφου σας. Ας περάσουμε τώρα στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης, το οποίο δεν βρίσκεται πολύ μακριά από αυτά τα οποία μόλις τώρα συζητούσαμε. Εξέταση λοιπόν του σχεδίου γνωμοδότησης όσον αφορά τις συμβάσεις για τη διαδικτυακή και άλλες εξαποστάσεως πωλήσει προϊόντων και το λόγο έχει καταρχάσει η κυρία Χάουταλα, η οποία είναι η συγκήτρια, συντάκτρα γνωμοδότησης. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Με ιδιαίτερη χαρά βλέπω ότι έχουμε όλους εδώ τους συγητές και συντάκτες γνωμοδότησης για τις δύο αυτές οδηγίες. Η μία έχει να κάνει με τις διαδικτυακές συμβάσεις όσον αφορά τα αυτά προϊόντα, ενώ η άλλη οδηγία έχει να κάνει με το λεγόμενο ψηφιακό άειλο περιεχόμενο. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που μπορούμε να συνεργαστούμε από κοινού προκειμένου να καταφέρουμε να ευθυγραμμίσουμε τις βασικές αρχές, τους βασικούς άξονες των δύο αυτών οδηγιών που έχουν να κάνουν τόσο με τους καταναλωτές όσο και με τους επιχειρηματίες και τους κατασκευαστές. Πρέπει βέβαια να σας πω ότι όσο περισσότερο μελετώ την επαναδιατύπωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τις συμβάσει πώληση ε, διαδικτυακών προϊόντων ή μάλλον τη διαδικτυακή πώληση προϊόντων, τόσο περισσότερο πείθομαι ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με το ζήτημα λίγο περισσότερο. Και ήδη φάνηκε από την προηγούμενη συζήτηση ότι οι διαδικτυακέ και μη διαδικτυακέ συμβάσει πώληση προϊόντων, και όταν λέμε μη διαδικτυακή εννοούμε κάθε μορφή πώληση που λαμβάνει η χώρα στην εσωτερική αγορά για τα υλικά προϊόντα, τότε στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να έχουμε απόλυτη εναρμόνιση για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Ο τρόπος όμως με τον οποίο ανέλαβε δράση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάνοντας δηλαδή συστάσεις, προκειμένου να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της πρότασης αυτής και να μην καλύπτει μόνο τις ε, διαδικτυακές συμβάσεις αλλά και τις μη διαδικτυακές συμβάσεις. Η προσέγγιση λοιπόν αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν βρίσκει σύμφωνη τη δική μας την Επιτροπή, η οποία μάχεται για την καλύτερη νομοθεσία, για το θετήν. Πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μία ολοκληρωμένη μελέτη αντικτύπου για το ζήτημα της επέκτασης του πεδίου εφαρμογή, γιατί θεωρούμε ότι δεν τηρείται εν προκειμένου και η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Για ένα τόσο ουσιαστικό ζήτημα, για μια τόσο θεμελιώδη τροποποίηση τελικά που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επέκταση του πεδίου εφαρμογή, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να εμπλέξουμε περισσότερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά να μην είναι ο μόνος παράγοντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια νομοθεσία η οποία δεν θα δημιουργεί δυσάρεσες εκπλήξεις για τον καταναλωτή ή για τον επιχειρηματία. Μια νομοθεσία η οποία δεν θα περιπλέκει τα πράγματα περισσότερο, μια νομοθεσία η οποία δεν θα προωθεί περαιτέρω τον κατακαιρματισμό της αγοράς. Τον βασικό αυτό στόχο τον συμμερίζεται και ο συνάδελφο Ράντεφ, αλλά και οι υπόλοιποι εισηγητέ και συντάκτε γνωμοδότηση. Ήρθε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου να απευθυνθούμε πλέον επισήμω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να πούμε στην Επιτροπή να κάνει τη δουλειά που θα έπρεπε να είχε κάνει εδώ και καιρό. Πέρα από αυτά, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε πώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιο συγκεκριμένα η δική μα Επιτροπή θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε αυτή την εργασία σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 55 του κανονισμού και ξέρουμε ότι ο κύριος Άριμοντ είναι ο, ο εισηγητής για την Επιτροπή ΙΜΚΟ. Νομίζω ότι ήδη συμφωνούμε για πολλά σημεία και με τους υπόλοιπους συναδέλφους που ασχολούνται με τη διαδικτυακή πώληση προϊόντων και με τις σχετικές συμβάσεις, καθώς επίσης και με την πρόταση που έχει να κάνει με το ψηφιακό περιεχόμενο. Νομίζω ότι πλέον όλοι συμφωνούμε ότι τα προϊόντα αυτά που έχουν έναν σωματωμένο ψηφιακό περιεχόμενο θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας κυρίως για την οδηγία εκείνη που έχει να κάνει με τις ε, ψηφιακές, ε, μάλλον διαδικτυακές συμβάσεις για τα προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου. Επ' αυτού συμφωνούμε όλοι. Υφίστανται επίσης ε, διαφορές ανάμεσα στα, διάφορα, στα δύο αυτά είδη προϊόντων. Από τη μια δηλαδή τα υλικά προϊόντα και από την άλλη το ψηφιακό περιεχόμενο. Όσον αφορά τις προτάσεις που έχουν να κάνουν με τα πτά τελικά προϊόντα, θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε να διαγράψουμε την ιεραρχία αυτή αποζημιώσεων που προβλέπεται ή νομική, αν θέλετε θεραπείας, ότι θα πρέπει δηλαδή αναγκαστικά οι καταναλωτές να ακολουθούν μία συγκεκριμένη σταδιακή προσέγγιση προκειμένου να καταφέρουν να πετύχουν αποκατάσταση ή αποζημίωση. Όσον αφορά τώρα τις ε, διαδιακτικές πωλήσει, προφανώς εδώ πέρα θα πρέπει να έχουμε εναρμόνιση, θα πρέπει να έχουμε μια καλώς λειτουργούσα ψηφιακή αγορά, αλλά από την άλλη αυτό δεν θα πρέπει να γίνει εις βάρος συγκεκριμένων και εκτιμένων δικαιωμάτων του καταναλωτή, που έχουν να κάνουν με τις περιόδους παραγραφής για παράδειγμα ή και με άλλα ζητήματα. Θα έλεγα λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε ένα κάποιο βαθμό ευελιξίας αυτή την προσέγγιση μέγιστης εναρμόνισης και αυτό διότι δεν θέλουμε να προκύψουν καταστάσεις όπου οι καταναλωτέ θα νιώθουν τελικά ότι μάλλον χάνουν στα δικαιώματά τους παρά κερδίσουν νέα δικαιώματα. Στα πλαίσια αυτής της όλης εργασίας θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να γενικεύσουμε τη χρήση συγκεκριμένων καινοτομιών που έχουν κάνει ορισμένα κράτη-μέλη όσον αφορά την εθνική τους νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών. Την εγγύηση όσον αφορά τα κρυμμένα ελαττώματα, το Βέλγιο και η Γαλλία έχουν πολύ καλά εθνικά συστήματα από αυτού. Θα μπορούσαμε λοιπόν αυτό να το συζητήσουμε περισσότερο μεταξύ μόνο. Για ποιο λόγο να μην ισχύει ένα τέτοιο κανόνα, ένα τέτοιο σύστημα για το σύνολο των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι έχω καλύψει τα πιο ουσιαστικά στοιχεία να ολοκληρώσω απλώ λέγοντα ότι ε, η οδηγία αυτή θεωρώ ότι θα είναι πιο πολύπλοκη από την ε, οδηγία την οποία επεξεργάζονται οι συνάδελφοι για το ψηφιακό περιεχόμενο. Γιατί αυτή τη στιγμή πραγματικά βαδίζουμε σε ένα ναρκοπαίδιο. Ξέρουμε ότι ε, οι παρελθούσες απόπειρες εναρμόνισης σχετική νομοθεσία δεν ευωδόθηκαν, οδήγησαν σε αποτυχία. Πρέπει λοιπόν να καταβάλουμε εκ νέου σημαντικές προσπάθειες και ελπίζω ότι έχουμε αντλήσει διδάγματα από τις παρελθούσες αποτυχίες. Τελευταία παρατήρηση. Μία από τις επιπτώσεις της επέκτασης ε, του ε, πεδίου εφαρμογή της εν λόγω οδηγία όσον αφορά τα απτά υλικά αυτά αγαθά, για να καλύπτονται όχι μόνο οι διαδικτυακές συμβάσεις, αλλά και οι μη διαδικτυακές, μη επιγραμμικές συμβάσεις, αυτό θα οδηγήσει σε ακύρωση μια βασική οδηγία για την προστασία των καταναλωτών από το 1999. Προφανώς αυτό θα αποτελέσει ε, μία από τις συνέπειες, αλλά δυστυχώς δεν έχει γίνει ακόμα μία αξιολόγηση αντικτύπου για την απουσία τελικά της οδηγίας αυτής, για το τι θα συμβεί να ακυρωθεί τελικά αυτή η οδηγία. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να ασχοληθούμε εκ νέου πολύ με την προτινόμενη αυτή επέκταση του πεδίου εφαρμογή. Δεν ξέρω αν ο κύριο Αρημών θέλει να πάρει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ τη συνάδελφο Χάουταλα. Εμείς στην Επιτροπή ΙΜΚΟ είμαστε απόλυτα πρόθυμοι να παρακολουθήσουμε αυτά που έχει να μας πει η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και να τα λάβουμε και υπόψη στη δική μας συζήτηση. Θεωρούμε ότι μπορούμε να βασιστούμε σε κάποιες βασικές αρχές Πρώτον, ότι θα πρέπει να ενοποιηθούν οι διατάξεις για το επιγραμμικό και μη επιγραμμικό ε, ε, εμπόριο ε, για να προστατεύσουμε και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Πρώτον, για να μπορούν τέτοιου είδους επιχειρήσεις να ιδρύονται και στη συνέχεια για να μπορούν να αναπτύσσονται. Γι' αυτόν το σκοπό απαιτείται ένα κοινό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο ώστε να μην, μπορεί, να μπορούν, να μην μπορούν μόνο οι μεγάλοι παίκτες να αντέξουν σε αυτόν τον ανταγωνισμό στην πανευρωπαϊκή αγορά. Γι' αυτό και θα πρέπει να θεσπιστούν κοινοί κανόνες για το online και το offline εμπόριο. Πώς θα γίνει αυτό ε, είναι ένα ερώτημα ανοιχτό το οποίο θα συζητήσουμε και στον, ε, στην Επιτροπή ΙΜΚΟ και έχουμε ζητήσει και από το σχετικό τμήμα πολιτικής του Κοινοβουλίου να μας ε, υποβάλει μια γνωμοδότηση. Και βεβαίως θα ακολουθήσουν και διάφορες αξιολογήσεις. Είπατε επίσης ότι συμφωνούμε όλοι ότι χρειαζόμαστε την καλύτερη δυνατή εναρμόνιση. Όχι απαραίτητα πλήρη βεβαίως εναρμόνιση, αλλά την καλύτερη δυνατή εναρμόνιση για να αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό της αγοράς. Είπατε όμως ότι αυτή η ε, εναρμόνιση θα πρέπει να είναι και εύρυθμη. Και αυτό είναι και το σημαντικότερο θα πρέπει δηλαδή να κάνουμε κάτι το οποίο θα εξασφαλίζει υψηλέ προδιαγραφέ για του καταναλωτέ, αλλά που ταυτόχρονα θα δίνει και τη δυνατότητα στι επιχειρήσει να λειτουργούν στην ενιαία αγορά. Άρα θα μην δημιουργήσουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα αποτρέπει ή θα εμποδίζει τι επιχειρήσει από το να ιδρύονται ή από το να αναπτύσσονται. ευρωπαϊκέ δηλαδή διασυνοριακές online πλατφόρμες αυτή τη στιγμή ε, ανέρχονται μόνο στο 4% του συνολικού ε, ψηφιακού, ε, της συνολικής ψηφιακής αγοράς. Το υπόλοιπο 96% αφορά εθνικές πλατφόρμες πώλησης. Και αυτό είναι μια μορφή καταστροφής. Θα πρέπει μέσω του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν πανευρωπαϊκές πλατφόρμες πώλησης Γι' αυτό ε, πιστεύω ότι χρειάζεται εναρμόνιση. Συμφωνώ με αυτό που είπατε ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί και μια κάποια ευελιξία. Αλλά αυτό είναι πάντοτε πολύ δύσκολο ως καθήκον. Το να θέλει δηλαδή κανείς να θεσπίσει μια νομοθετική διάταξη ή νομοθετικούς κανόνες και ταυτόχρονα να τους καταστήσει ευέλικτους. Αυτό για το βίσκασε που αναφέρατε εγώ είμαι ε, νομικός και ε, είμαι Βέλγος και έχω κληθεί στη ζωή μου να ε, χρησιμοποιήσω και να αξιοποιήσω αυτήν την διάταξη. Πρέπει όμως να σας πω ότι ο καταναλωτής πολλές φορές δεν γνωρίζει τα δικαιώματα του. Γνωρίζει τα δύο χρόνια της εγγύησης, αλλά δεν γνωρίζει το ζήτημα αυτό του, του βίσκασε, του κρυμμένου δηλαδή ελαττώματος. Ε, αυτό που θα πρέπει ενδεχομένως λοιπόν να εξετάσουμε είναι ε, ε, ε, μήπως θα έπρεπε να θεσπιστεί μια τέτοια ε, ρύθμιση χωρίς να καταργείται αυτό το, αυτή η διάταξη, αυτός ο κανόνας του Βίσκασε που αναφέρατε. Αυτό ήταν το πρώτο. Το δεύτερο που θα ήθελα να αναφέρω σχετίζεται με το lifespan, με τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Το, συζητήσαμε και στο προηγούμενο θέμα. Ε, και εδώ ίσως θα μπορούσα να ε, προτείνω αυτό που πρότεινε ο κύριος Τόνερ. Μήπως θα έπρεπε δηλαδή το ζήτημα αυτό να ρυθμίζεται σε επίπεδο κατασκευαστή. Τώρα, αν τα δύο συν δύο χρόνια που αναφέρονται στην έκθεση, τα, δύο χρόνια εγγύηση συν δύο χρόνια ε, αντιστροφής του βάρους απόδειξης, θα πρότεινα να αποφύγουμε μια τέτοια λύση, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι όλοι όσοι ε, δραστηριοποιούνται στην αγορά να έχουν εμπιστοσύνη σε αυτήν. Και με αυτόν τον τρόπο ε, Αντιθέτω, ε, επιτυχάνεται το αντίθετο αποτέλεσμα. Γιατί σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει κάθε φορά κάποιο κατασκευαστή προϊόντο να εξετάζει με το νομικό του τμήμα τη εταιρεία του αν έχει το δικαίωμα να πουλήσει το τάδε προϊόν στην Πορτογαλία ή στη Φιλανδία κτλ. κτλ. Πάντως σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σα και σα διαβεβαιώ ότι θα τα λάβω υπόψη μου και στην περαιτέρω δουλειά μου. Ε, η κυρία Γκέπχαρτ, ευχαριστώ. Είμαι η ε, σκιώδη συγκίτρια των σοσιαλιστών. Ε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την κυρία Χάουτελα για την εξαιρετική ε, έκθεσή της που, με την οποία συμφωνώ ε, στα περισσότερα σημεία και την οποία αποδέχομαι. Θα ήθελα ωστόσο να επισημάνω ένα θέμα στο οποίο δεν συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Χάουτελα ακριβώς γιατί γι' αυτό το λόγο κάνουμε και αυτή τη συζήτηση. Μιλώ για τους ορισμούς. Είχαμε συμφωνήσει, Ίμκο και Γιούρι, οι ορισμοί εκείνων που, των ε, όρων που ε, εμπίπτουν στο πεδίο ισχύω, ε, στο στην οδηγία για τα online προϊόντα και για τα υλικά προϊόντα να μην παρουσιάζουν διαφορές. Στην τροπολογία 3, ωστόσο, εσείς θέλετε να υπάρξουν αλλαγές ε, σε ορισμένα προϊόντα και να, αφαιρέσουν, να, να αφαιρεθούν για παράδειγμα τα USB, τα CD και τα DVD. Ώστε αυτό όμως θα έχει ως αποτέλεσμα να μην αναφέρονται αυτά τα προϊόντα ε, σε, καμία, σε κανένα νομοθέτημα. Πράγματι θέλατε να δημιουργήσετε αυτό το κενό ή μήπως θα ήταν καλύτερο να ε, δημιουργήσουμε ένα τέτοιον ορισμό που θα καλύπτει όλα τα είδη προϊόντων Αυτό θα με ενδιέφερε πολύ, πρέπει να σας πω. Σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογής, offline και online, εδώ τα πράγματα είναι σαφή, πραγματικά δεν μπορεί να υπάρχει διάκραση, δεν μπορεί να έχουμε διαφορετικό δίκαιο αναλόγως του αν αγόρασα κάτι στο, σε ένα κατάστημα ή στο ίντερνετ, είναι πραγματικά παράλογο κάτι τέτοιο και γι' αυτόν τον λόγο ε, σας υποστηρίζω πλήρως ως προς αυτό. Σε ό,τι αφορά την, ε, το ζήτημα των ε, δικαιωμάτων εγγύησης ε, συμφωνώ μαζί σας, μέχρι στιγμής υπάρχει ελάχιστη εναρμόνιση δύο χρόνια. Σε κάποιες χώρες ισχύουν μεγαλύτερες προθεσμίες, δύο, τρία έτη. Ε, σε κάποιες χώρες προβλέπεται η διάρκεια ζωής του προϊόντος. Όλα αυτά είναι ζητήματα, είναι, είναι εργαλεία ευελιξίας, τα οποία δεν, πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να τα χάσουμε. Γιατί λοιπόν οι καταναλωτές να χάσουν αυτά τα δικαιώματα που τα απολαμβάνουν ήδη. Ε, πρέπει δεν να σας πω ότι και μια ε, Πολωνή η οποία ε, αγοράζει online ένα προϊόν από τη Γαλλία καλύπτεται και εκείνη από τα τρία χρόνια της εγγύησης. Άρα θα πρέπει η νομοθεσία να συμβάλλει στην ενίσχυση και στη διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου. Και όσον αφορά την ιεράρχηση των δικαιωμάτων δηλαδή επιδιόρθωση ή αντικατάσταση και αυτό το θέμα θα χανόταν από μια εναρμόνιση ε, στις χώρες όπου ήδη προβλέπεται κάτι τέτοιο. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι η πλήρης εναρμόνιση είναι πάρα πολύ προβληματική εκτός εάν ο πύχης τεθεί πάρα πολύ ψηλά. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσα να συμφωνήσω και εγώ με την πλήρη εναρμόνιση, αλλά όπως είπα θα πρέπει πραγματικά να ε, τεθεί πάρα πολύ ψηλά ο πύχης. Όσον αφορά την αντιστροφή του βάρους απόδειξης μίλησα νωρίτερα και για το Βισκασέ πρέπει να σας πω ότι είναι ένα ζήτημα που με απασχολεί και εμένα, κάτι που υπάρχει δηλαδή στη Γαλλία και στο Βέλγιο και δεν είναι σαφές μήπως ε, μέσω μιας πλήρους εναρμόνισης αυτοί οι σχετικοί κανόνες καταργούνταν στις χώρες όπου ισχύουν. Ξέρω ότι ε, οι κανόνες αυτοί δεν είναι πάντοτε γνωστοί σε όλους τους πολίτες, αλλά όποτε ε, επισημαίνεται σε κάποιον πολίτη ότι έχει αυτό το δικαίωμα, τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ θετικά. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά σε περίπτωση ε, μήπως μάλλον ε, αν προσπαθήσουμε να καταργήσουμε καταναλωτικά δικαιώματα τα οποία ισχύουν ήδη σε κάποιες χώρες, μήπως τροφοδοτούμε τους ε, ακροδεξιούς και τους λαϊκιστές οι οποίοι θα βγουν και θα πούν ότι να δείτε τι κάνει η Ευρώπη Μήπως είναι και αυτά όμως εμ, διαστάσεις τις οποίες θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, να είμαστε πάρα πολύ ε, προσεκτικοί ε, ως προς την πρόταση που θα καταθέσουμε ε, και τις, ε, το, το δικό μας σκεπτικά. Γι' αυτό εμείς ως σοσιαλδημοκράτες πρέπει να σας πω ότι με αυτή την προσέγγιση δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα. Σχετικά με το η χώρα μου όπως και άλλες έχουν μακρά ιστορία ε, στηρίζουν αυτή την πρακτική και τις ε, εκθέσεις ε, περί αξιοπιστίας τώρα, αλλά οι οργανώσεις καταναλωτών τόνισαν ότι αυτή η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται μετά από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους και σωστή λογοδοσία. Και θα πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που με απασχολεί σχετικά με αυτή την πρόταση. Κάτω πρόσδεκτη η πρότασή σας, συμφωνούμε με τα ένδικα μέτρα τα οποία προτείνετε, τον τρόπο θεραπείας. Πιστεύω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να κοιτάξουμε προκειμένου τα δικαιώματα του καταναλωτή να μην ε, επηρεάζονται αδίκως. Τώρα το άρθρο 17 σχετικά με την Νομίζω ότι αυτό το συγκεκριμένο άρθρο είναι πολύ αδύναμα διατυπωμένο σε ό,τι φορά το ψηφιακό έντυπο. Ψηφιακό περιεχόμενο, συγγνώμη. και το ζήτημα του σεβασμού της οδηγίας δεν ε, εκφράζεται με τρόπο ιδιαίτερα ρητό. Από την εμπειρία μου, ε, οι διατάξεις περί επιβολής θα έπρεπε να είναι πολύ πιο στεναρά διατυπωμένες τέσσερα στα πρώτα μέλη να μην έχουν ε, τη δυνατότητα να τις παρακάπτουν. Θα το συζητήσουμε σε δυο μας περαιτέρω. Ο κύριος Στάντ Μάιερ, εκ μέρους της Κομισιόν, θέλει να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια ζωής, που ήταν το προηγούμενο σημείο, αλλά επανέρχεται εδώ. Κύριε Χάουταλα αναφέρθηκε στους πόρους και την ανάγκη ε, λήψη υπόψη τη διάρκεια του προϊόντος. Ε, φυσικά, η Κομισιόν συμφωνεί απόλυτα ανέλησε η Κομισιόν το ζήτημα και ταυτόχρονα ε, προτείναμε το πρόγραμμα για την κυκλική οικονομία. Το θέμα είναι αυτό που περιλαμβάνεται στο εκτιμώντας 23. Να εξηγήσω λίγο πιο ουσιαστικά το θέμα. Κατανοούμε απόλυτα τα επιχειρήματα για συμπέρληψη κριτηρίων ε, διάρκεια ζωής και της συμμόρφωσης, αλλά ε, προκύπτει πρόβλημα εάν ξεπεράσουμε την προθεσμία για την, τις εγγύησεις, δηλαδή τη διετία. Για ποιο λόγο, υπάρχουν δύο διαφορετικά συστήματα που λοιπόν, διαφορετικό χαρακτήρα. Ε, έχετε τους, ε, τε, ε, τους κανόνες ή αν ε, ακολουθήσουμε την άποψη του κ. μας, τότε υπεύθυνο είναι ο, καταναλω... ο κατασκευαστής. Αυτή είναι η πρώτη διαφορά. Η δεύτερη διαφορά είναι ότι οι πωλήσει αφορούν όλα τα προϊόντα. Μια τεράστια ποικιλία. Και γι' αυτό θα πρέπει να είναι απλές και να παρέχουν νομική ασφάλεια. Όπως εξήγησε και στο Τόνερ, δεν πρόκειται για τεχνικά προϊόντα ή άρα προϊόντα ε, διαρκείας ε, όπως τα έπιπλα και η τρίτη διαφορά, ε, ε, πιο σημαντική, είναι ε, αφορά την προθεσμία, τη διάρκεια λήξης. Προτείνεται διετής περίοδος, αλλά θα πρέπει, κατά την άποψή μου, να υπάρχει μία περίοδος για όλα τα προϊόντα. Όλα τα αντιμετωπίζουμε με τον αυτό τρόπο, από χρονική σκοπιά. Τώρα, η διάρκεια του προϊόντος είναι άλλο πράγμα και ο κύριος Τόνερ εξήγησε ότι το κριτήριο το οποίο συνδέεται με την ένταση και τη συχνότητα χρήσης του προϊόντος ε, παίζει ιδιαίτερη σημασία παρά ένα χρονικό περιθώριο. Αν πάρετε μια ηλεκτρική σκούπα και αναφέρετε 5.000 ώρες ε, χρήσης, είναι διαφορετικό αν κάποιος το χρησιμοποιεί μία ώρα την εβδομάδα ή πολλές ώρες την ημέρα. Αν το χρησιμοποιείς ε, κάθε μέρα με εντατικό τρόπο, τότε φτάνεται στον όριο ζωής, διάρκεια ζωής πολύ πιο γρήγορο. Εδώ αυτό λοιπόν όταν εστιάζουμε στο, θέμα της διάρκειας ζωής θα πρέπει να εστιάσουμε ιδιαίτερα στην ένταση και την ε, συχνότητα της καθίσης. Η Κομισιόν ανέλησε το Ολλανδικό σύστημα και έκανε την πρόταση διότι η Ολλανδία έχει ένα σύστημα το οποίο βασίζεται στη διάρκεια της ζωής <clears throat> και μετά αυτό αφορά διάφορες περιόδους. Φυσικά εδώ έχουμε ένα πίνακα που έχει συντάξει ο κλάδος ε, για ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά αγαθά. Είναι μια συμφωνία που έχουν συνάψει όλοι οι βιομήχανοι του κλάδου έχουν φτιάξει 10 υποκατηγορίες για τηλεόραση, φορτά τηλέφωνα, υπολογιστές, μηχανές καφέ κλπ. 10 διαφορετικές υποκατηγορίες και σε κάθε υποκατηγορία υπάρχει υπο-υποκατηγορία ανάλογα με την τιμή. Από μία κατηγορία έως 7 διαφορετικές υποκατηγορίες και το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχουν 29 διαφορετικές περίοδοι. 29 διαφορετικές περίοδοι. Και όταν κάναμε την άσκηση REFIT, ζητήσαμε από όλους τους εμπλεκόμενους και όλοι συμφώνησαν ότι αυτό δεν είναι ένα σύστημα που δίνει νομική ε, ασφάλεια δικαίου. Για ε, νόμο περιπολίσεων πρέπει να έχετε μία περίοδο, η διάρκεια δεν έχει τόση σημασία, αλλά είναι μία μοναδική περίοδος. Εάν μιλάτε τώρα για ε, μη αναλώσιμα προϊόντα διάρκειας, αγαθά διαρκείας, τότε αυτό βασίζεται και σε το θέμα της, των διαφορετικών κριτηρίων συμμόρφωσης. Και για να απαντήσω ακόμα, δεν θέλω, κάτι, σε κάτι ακόμα, δεν έχω χρόνο, σε αυτό που είπε η κυρία Χάουταλα για την μελέτη δικτύπου. Είναι πολύ ενδιαφέρον να υποβάλλονται προτάσεις που έχουν ε, στοιχεία αλλά εμείς ε, σας παρήχαμε τα στοιχεία τον, ε, τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο και μπορούμε να πάει στιγμή να σας ε, υποβάλουμε περαιτέρω στοιχεία. Το τρίτο στοιχείο που θα ήθελα να αναφέρω είναι η πλήρης εναρμόνιση. Είναι ιδιαίτερη σημασία. Δεν θα ήθελα να επισέλθω σε λεπτομέρειες, απλά να τονίσω ένα σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, το συμφέρον των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων. Και ποιο είναι το συμφέρον των επιχειρήσεων. Είναι η πλήρης εναρμόνιση. Δεν είναι ζήτημα που βάζουμε τον πύχη σε ρουφά την προσθέτει του καταναλωτή. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα μόνο ε, σύνολο κανόνων Εάν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, τότε δεν ε, έχει ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις ένας τέτοιος κανόνας. Γι' αυτό λοιπόν, εάν σε διάφορα κλάστερ, όπως είπε και η κυρία Χάουταλα, ένα σύστημα που θα πηγαίνει υψηλότερα, τώρα όλα τα βασικά κλάστερ της Κομισιόν, όπως το θέμα της ιεράρχησης, ε, όχι να είναι διετή περίοδο αλλά να βασίζεται στην διάρκεια ζωή σε ένα κρυφό ελάττωμα και το θέμα της αντιστροφή του βάρους αποδείξης, όλα αυτά είναι τέσσερα σημεία, τα οποία είναι τα βασικά σημεία αυτή της προτάσεως και επίσης να πω ότι μπορεί να έχουν τους ίδιους κανόνες, αλλά, αλλά όχι. Τώρα ας μπούμε στη θέση ε, κάποιου ο οποίος θέλει να πωλήσει, να τα προϊόντα του στην Ευρώπη. Νομίζω πως ε, αν προέρχεται εκτό Ευρώπη δεν θα το επιδιώξει. Θα πρέπει να συνεργαστούμε και να συζητήσουμε με το Κοινοβούλιο ως Κομισιόν. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, Ευχαριστούμε. Επρόκειτο για την τελευταία παρέμβαση για το σημείο αυτό. Να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι η 10η Ιανουαρίου. Περνάμε στο επόμενο σημείο της μέρας της διάταξης, το οποίο θα εξεταστεί και κλεισμένο των θυρών Όσοι δεν έχουν το δικαίωμα πλέον να παραμείνουν στην αίθουσα, σας παρακαλώ πολύ να αποχωρήσετε. Κύριε Τόνερ, κύριε καθηγητά Τόνερ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα.